κάνουμε κάτι τέτοιο κατά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας, κατά τη σύνοδο. Ε, πρέπει να ομολογήσω ότι η έλλειψη ομοφανίας σχετικά με τις συγκεκριμένες αποφάσεις μπορεί να θεωρηθούν ως οπισθοχώρηση στην πολιτική μας στα Δυτικά Βαλκάνια και την πολιτική διεύρυνση που παραμένει στρατηγική επένδυση ε, για την σταθερότητα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτό σίγουρα δεν σημαίνει όμως ότι θα σταματήσουμε εδώ. Σημαίνει μόνο ότι ακόμα περισσότερες προσπάθειες είναι απαραίτητες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις στο Συμβούλιο σε σχέση με τη δέσμευσή μας υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Η σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης μάλιστα της εμπλοκής της Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια είναι κοινή ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι επίσης σαφές ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ότι η περιοχή είναι στην αυλή μας και πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους βοηθήσουμε στις μεταρρυθμιστικές τους διαδικασίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε μια μακρά συζήτηση την περασμένη εβδομάδα για αυτό το θέμα και στο τέλος οι ηγέτες συμφώνησαν να επανέλθουν στο θέμα αυτό πριν από τη Σύνοδο στο Ζάγκρεμπ το Μάιο του 2020. Στο Συμβούλιο είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ε, ό,τι χρειάζεται. Η Προεδρία παραμένει δεσμευμένη να κάνει αυτό που μπορεί, ούτως ώστε να διερευνήσει μια οδό προς ένα σαφές και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να επαναλάβω επίσης πόσο σημαντικό είναι και η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία να συνεχίσουν να κάνουν συγκεκριμένες προόδους στις μεταρρυθμίσεις. Αυτό χρειάζεται για την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πιο σημαντικό πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται οι λαοί και των δύο αυτών χωρών. Επίσης, είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η δέσμευση υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών παραμένει σημαντική για όλα τα, μέλη, για όλα τα μέρη που επιθυμούν ένταξη. Τέλος, να ε, εκφράσω την εκτίμησή μας προς τη Βόρεια Μακεδονία ε, για το θάρρος της να ε, προχωρήσει στη Συμφωνία των Πρεσπών και την αλλαγή του ονόματος. Επίσης, χαιρετίζομαι την πολιτική βούληση να προχωρήσουν που ε, ε, έδειξε πάντοτε η κυβέρνηση στην Αλβανία παρά την πόλωση στο πολιτικό κλίμα. Είμαι πεπισμένος ότι σύντομα θα έρθει η ώρα να ανταμυφθούν οι προσπάθειες αυτές. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Minister. Now, on behalf of the Commission... ευχαριστούμε τώρα ε, και, τώρα εκ μέρους της Επιτροπής ο, κύριος Χάν έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αυτό το οποίο έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αστόχησαν να εκπληρώσουν τις εξαγγελίες τους όσον αφορά την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν να δίνουν το πράσινο φως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά δυστυχώς δεν ήταν όλες οι χώρες μέλη έτοιμες να πάρουν αυτή την απόφαση. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στην κυρία Ράινεν για την προσωπική της βούληση και τις ε, προσπάθειες για την εξέβρεση μιας λύσης μερικές μέρες ε, πριν στο ε, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Αυτό δεν έγινε δυνατό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να υποφελθώ της παρουσίας των μελών του Συμβουλίου για να τα ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κατέβαλαν με το επιτελείο τους. Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατό να εξεύρουμε μια συμφωνία ε, προκάλεσε στήματα βαθιά απογοήτευση. Αυτό το, θα ήθελα να παραλάβω αυτό το που είπα την περασμένη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο. Δεν πρόκειται για μια στιγμή θριάμβου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Και ας μην λησμονούμε ότι υπάρχει ομοφωνία για ένα πράγμα. Τα Δυτικά Βαλκάνια χρειάζονται πολύ περισσότερες ε, θαραλές αποφάσεις. Μετά από την αποτυχία μας αυτή θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα απαντήσουμε τα εξής ε, ερωτήματα Πού βρίσκονται οι δεσμεύσεις μας και η υποστήριξη προς εκείνους που πήραν τα σημαντικά πολιτικά ρίσκα. Χρωστάμε στις χώρες, ε, το λιγότερο που χρωστάμε στις χώρες Βαλκανικής είναι εντιμότητα. Η διεύρυνση δεν σημαίνει ότι είμαστε καλοί με τους γειτονές μας. Ε, σημαίνει, ότι ε, ερχόμαστε, προσερχόμαστε έγκυρα στο ραντεβού μας με την ιστορία οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη θα πρέπει τώρα να διευκρινίσουν πόσο σοβαρή είναι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης όσον την ένταξη αυτών των χωρών. Δεν θα πρέπει να κατηγορήσουμε ούτε τη Βόρεια Μακεδονία ούτε την Αλβανία για την αποτυχία. Και δύο χώρες εκπλήρωσαν τα όσα του ζητήσαμε και ακόμα και περισσότερα πράγματα και το αναγνωρίζουν ε, και οι σχετικές εκθέσεις. Έγιναν σημαντικές πρόοδοι όσον αφορά το κράτος δικαίου, δικαστική μεταρρύθμιση, πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου, οργανωμένου εγκλήματος. Ε, επιπλέον, η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν πραγματικά ένα εξαίρετο επίτευγμα, το οποίο βασίζεται στο σθένος και την ε, αποφασιστικότητα να ξεπεραστούν τα εμπόδια χάρη ενός ευρύτερου μέλλοντος για τις δύο χώρες. Η ευθύνη μας τώρα είναι να ε, σταθούμε στο πλευρό των χωρών αυτών, των οποίων οι πολίτε αισθάνονται βαθιά απογοητευμένοι. Δεν θα πρέπει να παραιτηθούμε από όλε τι ελπίδε μα. Η δέσμευσή μα ε, όσον αφορά την προοπτική τη ε, ένταξη των χωρών τη Βαλκανική στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει. Γιατί η περιοχή αυτή παραμένει ένας, ένας πολιτικά στρατηγικός μας στόχος και αυτό προς όφελος και των δύο πλευρών. Γι' αυτό ε, θα συνέλθει η Σύνοδος Κορυφής το Μάιο του 2020 στο Ζάγκρεπ και ελπίζω να υπάρξει τότε μια θετική έκβαση. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία με κάθε τρόπο που μπορεί, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται προς όφελος των πολιτών αυτών των χωρών ε, προκειμένου να τις καλωσορίσουμε μελλοντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να σταθούμε στο πλευρό των πολιτών αυτών των χωρών και της ευρύτερης περιοχής. Κατανοώ πλήρως ότι η αποτυχία αυτή ε, προκάλεσε μια τεράστια απογοήτευση. Παρόλα αυτά, ε, θα πρέπει να παράσχουμε τη δική μας συνδρομή προκειμένου να ξεπεραστεί η κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα θα ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών. Εκ μέρους του ΕΛΚ έχουμε ως πρώτο ομιλητή τον κύριο Κόβατσεκ. E Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι απογοητευμένο από την ανικανότητα του Συμβουλίου να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις δύο αυτές χώρες. Το μήνυμα του Συμβουλίου στέλνει ένα απέσιο γεωπολιτικό μήνυμα ενάντια με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Στα πλαίσια της συνάντησης κορυφής του Ζάγκρεπ θα πρέπει να επανορθώσουμε το λάθος αυτό. Το μπλοκάρισμα αυτό θα έχει πολιτικές συνέπειες όχι μόνο στις δύο χώρες αλλά στο σύνολο της περιοχής. Η Βουλγαρική Προεδρία έθεσε το θέμα της διεύρυνσης 15 χρόνια μετά από τη συνάντηση κορυφής της Θεσσαλονίκης. Είναι προς το συμφέρον μας ε, να προχωρήσουμε στην ενσωμάτωση των χωρών αυτών. Άλλοι γεωπολιτικοί παίκτες όπως η Ρωσία, ε, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες ε, θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν βάρος στην περιοχή. Πρέπει επίσης να επενδύσουμε αρκετά σε ε, κατάλληλα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την προπαγάνδα εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές. Υπάρχουν πολλά που μένει να γίνουν όπως η Συμφωνία Καλής Γειτονίας ανάμεσα στη Σόφια και τα Σκόπια δεν έχει προχωρήσει. Διαρωτώ με γιατί μόνο ε, κάτω από πίεση από το εξωτερικό οι χώρες μπορούν να ξεπεράσουν τέτοιου είδους ε, συκοφαντικές ερμηνείες του ιστορικού τους παρελθόντος. Εν πάση περιπτώσει η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να εξαρτάται από την ικανότητα ενός ε, πολιτικού ηγέτη και ενός άλλου να καταστρέφει τις συμφωνίες αυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει οι χώρες του Συμβουλίου να μην μπλοκάρουν πλέον τις διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν οι διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία που θα χρειαστούν πολύ χρόνο έτσι κι αλλιώς για να ανακτήσουμε ταχύτατα την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κόβατσεφ, δέχεστε μία μπλε κάρτα. Κανονικά, κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των ομιλητών δεν δεχόμαστε μπλε κάρτα. Συνεπώς δεν μπορώ να δεχτώ το έτοιμά σας. Περνάω στον επόμενο ομιλητή, την κυρία Πύρη, για 1,5 λεπτό από πλευράς των Σοσιαλδημοκρατών. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Σακύρη, τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βόρειας Μακεδονίας. Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία αχ, υπόθηκε πέρυσι ότι έκαναν τις δύσκολες αλλά απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και γι' αυτό τους δώσαμε συγκεκριμένες υποσχέσεις και θα έπρεπε λοιπόν με τη σειρά της Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Η Βόρεια Μακεδονία είναι υποψηφία για 14 χρόνια και πήρε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια. Τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με το όνομα της χώρας οδήγησαν στην ιστορική συμφωνία των Πρεσπών και χρειάστηκε πολιτικό θάρρος ε, για να υπάρξει και από πλευράς Ελλάδας και από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας ένα τέλος στην ιστορία αυτή θάρρος. Το θάρρος που δεν είχαν όμως οι ηγέτες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το πω ή ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας δεν είχε. Ο κύριος Μακρόν δεν επέδειξε το πολιτικό θάρρο που απαιτείται από ένα ηγέτη. Δεν μπόρεσε να έχει την οριμότητα και την στρατηγική δυνότητα που απαιτείται από ένα ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλές φορές ε, υψώνει τη φωνή της σε θέματα στα οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε και πολύ τα πράγματα. Και το Συμβούλιο τελικά ήταν πολύ σιωπηλό σε σχέση με μια πολιτική επιλογή την οποία μπορούσαμε να επηρεάζαμε. Λυπάμαι, αλλά η συνάντηση κορυφή στο Ζάγκραπ το 2020 τον Μάιο είναι πολύ αργά, έρχεται πολύ αργά. New Europe Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ε, παρά τη μεγάλη υποστήριξη για τρίτη φορά σε ε, έξι μήνες το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να αρχίσει διαπραγματεύσεις. Πολύ απογοητευτική απόφαση με πολλές συνέπειες ενό ίσως ιστορικού λάθους. Δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που είχαμε υποσχεθεί πολλές φορές. Και αυτή η καθυστέρηση υποσκάπτει την ευρωπαϊκή αξιοπιστία στην περιοχή. Μετά, τη... Μετά από αυτή την ε, έλλειψη απόφασης ε, προκυρήθηκαν πρόορες εκλογές ε, ο ε, Πρωθυπουργό ήταν μεγάλος ε, σύμμαχο μας στην περιοχή. Η Βόρεια Μαχεδονία και η Αλβανία συνεχώ απέδειξαν ότι ανταποκρίνονταν έγκαιρα, κυρίω και στην κρίση με του πρόσφυγε και πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει. Θα πρέπει επί της αρχής των ιδίων αξιών να αξιολογηθούν οι χώρες αυτές. Εγώ προέρχομαι από χώρα που έπρεπε να περάξει να περάσει πρόσφατα από ενταξιακέ διαπραγματεύσει, γνωρίζω ότι η διαδικασία είναι γραφειοκρατική και στηρίζεται σε νομικέ διατάξει. Καμιά φορά όμω. Ε, ε, ε, αυτό δεν αρκεί. Ε, θα πρέπει να ε, δράσουμε έγκαιρα πριν από το Μάιο και το σύνοδο του Ζάγκρεμ. Αλλιώς υπονομεύομαι το όνειρο των ε, χωρών αυτών να προσχωρήσουν στην Ευρώπη και δημιουργείται ε, απογοήτευση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιουτικόφερ, δύο λεπτά από τους Πρασίνους. Κυρία Πρόεδρε, ένας πολύ γνωστός Γάλλος ε, σχολίασε κάποιες πολιτικές αποφάσεις ως εξής. Είναι χειρότερες από έγκλημα. Είναι λάθος. Η απόφαση του Συμβουλίου να αρνηθεί την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων είναι λάθος ιστορικών διαστάσεων. Ευχαριστώ τους ε, κυρίους Τούσκ, Γιούνκερ, Χάν, την κυρία Τούπουράινεν και όλους τους άλλους συναδέλφους που επέκριναν σαφώς την απόφαση αυτή του Συμβουλίου. Παρά την ε, οργή ε, μετά από το γεγονός ότι δεν τήρησε τις ε, ε, υποσχέσεις της, παρά τη μειοπική πολιτική, παρά την απογοήτευση που προκάλεσε στους λαούς της Μακεδονίας και της, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, αυτά ε, δεν θα τα αναφέρω, θα απευθυνθώ στον πρόεδρο Μακρόν. Κύριε Πρόεδρε, ε, σε αυτό το θέμα είστε απομονωμένος, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να ρίξει γέφυρα προς εσάς. Αν διαβάσετε προσεκτικά το ψήφισμά μας θα διαπιστώσετε ότι είμαστε διατεθειμένοι να ε, συμμετάσχουμε στις ε, ε, διαπραγματεύσεις για την μεταρρύθμιση της ενταξιακής διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει να συνεργαστούμε, αλλά διορθώστε το λάθος που εκάνατε. Δεν πρέπει να μείνουν στο κατόφλι Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία επειδή εμείς δεν κάναμε την δουλειά που έπρεπε στα του οίκου μας. Ευχαριστώ από την ομάδα ID η κυρία Άννα Μπονφρίσκο. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Όλοι γνωρίζουμε τις βαθύτατες πληγές που ε, έχει η περιοχή αυτή και που απειλούν Ξέρουμε την επιρροή της Κίνας, την επιρροή της Ρωσίας, την παρουσία ε, εγκληματικών δικτύων, τρομοκρατικών, ολιγαρχικών καθεστώτων, ε, παρέμβαση ε, των Τούρκων, πάνω από 50% μουσουλμάνοι στην Βοσνία και την Αλβανία, 28% στη Βόρεια Μακεδονία, και αντίστοιχα ποσοστά στο κοσυφοπαίδιο. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Χάν, μια σωστή εμπορική πολιτική από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να ακολουθηθεί ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι μια κοινή εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να θέσουμε σε δοκιμασία πάλι τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Τα συμφέροντά τους είναι το πιο σημαντικό για μας. Εξ ονόματος των Ευρωπαίων Συντηρητικών, η κυρία Φώτιγκα. Εδώ και πέντε χρόνια ε, στη δήλωση του κυρίου Γιούνκερ για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε μια σημαντική κρίση με τις σχέσεις μας ε, ε, με τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίτροπε, γνωρίζετε τι μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται από πλευρά σας, από πλευρά του προσωπικού σας, από πλευρά των Ευρωβουλευτών και των πολιτικών ηγετών να αναστραφεί ένα αρνητικό κλίμα. Και οι δύο αυτές χώρες, και η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία, ε, αξίζουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, έχουν εκπληρώσει αν πολλής, ε, τα κριτήρια τα οποία απαιτούνται μετά από πάρα πολλά χρόνια αναμονής. Και τώρα ξαφνικά έρχεται ένα χαστούκι από το Συμβούλιο. Ε, καταλαβαίνω το τι συμβαίνει σε διάφορες ε, χώρες όπως τη Γαλλία με τη στήριξη της Δανίας και της Ολλανδίας δημιούργησαν μια νέα κρίση στις σχέσεις μας με τα Δυτικά Βαλκάνια. Η κρίση αυτή θα αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη. Γι' αυτό λοιπόν η απόφαση του Συμβουλίου θα πρέπει να ακυρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Φτάνουμε τώρα στην Ενωμένη ε, Ευρωπαϊκή Αριστερά. 1,5 λεπτό ο κύριος Κούλογλου. Ξέρετε, τα δυτικά Βαλκάνια είναι η πιο ευάλωτη περιοχή στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι ε, συγκροτήθηκαν ε, μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το κομμάτι της ευρωπαϊκής μας ιστορίας. Ε, πρόσφατα η Βόρεια Μακεδονία έκανε ένα σημαντικό βήμα. Μαζί με την ελληνική κυβέρνηση ε, συνήψαν την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών ε, σε πείσμα του εθνικισμού και, ε, και του λαϊκισμού. Και τώρα, αντί να συνδράμουμε τον κύριο Ζάεφ, τον ε, οθούμε σε μια πολιτική αναταραχή. Γιατί αντί να εξαγάγουμε τις ευρωπαϊκές ιδέες της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης, εξάγουμε τα εσωτερικά μας πολιτικά προβλήματα. Και υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο θα έπρεπε να διατυπώσουμε προς τους κυρίους αυτούς. Ε, καταρχήν θα πρέπει να είναι παρόντες σε αυτή τη συζήτηση. Δεύτερον, δεν θα, πρέπει, θα πρέπει να σταματήσουν να παίζουν ε, μικροπολιτικά παιχνίδια με αυτές τις μικρές χώρες οι οποίες χρειάζονται την βοήθειά μας. Γιατί ακριβώς είναι μοιρέ, ε, μικρές και πρόσφατα συσταθήσεις. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Καστάλντο δεν παρίσταται όμως, γι' αυτό θα περάσουμε στην κυρία Ζόφκο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε Ε, ήθελε να υποστηρίξει τις χώρες αυτές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εγώ είμαι ε, βαθιά απογοητευμένος μετά όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα, γιατί οι χώρες αυτές εργάστηκαν σκληρά προκειμένου να πετύχουν τις δεσμεύσεις τους και να εκπληρώσουν τα κριτήρια για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ε, όλοι ελπίζαμε ότι οι προσπάθειές τους θα επιβραβευθούν με θετικά μηνύματα. Αντί γι' αυτό πήραν, ένα χαστούκι στο κατά πρόσωπα. Οι δύο αυτές ε, χώρες ε, χρειάστηκε πολλές φορές να απορρίψουν ελκυστικά και προσφορές από άλλες ε, περιοχές. Με τον τρόπο αυτό δίδεται ευκαιρία σε άλλους ε, παίκτες να εισχωρήσουν στο κενό που άφησε πίσω της η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνιστά μείζον στρατηγικό σφάλμα και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, την υπονομεύει. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Επίτροπο κ. Χάν για τις προσπάθειες τους. Δυστυχώς τα μέλη του Συμβουλίου ε, έδειξαν μια κοντόφθαλμη ε, στάση. Ε, μη ολοκληρωνεις μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από τον Ζακ Σιράκ. Η Προεδρία της Κροατίας έδειξε ότι το διακύβευμα είναι η ειρήνευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Πιτσούλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία κατάληξαν σε ένα ιστορικό σφάλμα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι πλοκαρίστηκε η πρόοδο λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων σε, μεταξύ κάποιων μελών ιδιαίτερα εκείνων που παρδόξου λένε ότι θέλουν να ανανεώσουν την Ευρώπη. Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία εκπλήρωσαν τους όρους που θέσαμε. Είναι απίστευτο το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει πολιτικό θάρρος έναντι της Βόρειας Μακεδονίας η οποία κατόρθωσε να επιλύσει τα προβλήματα που είχε με την ε, ε, γειτονά χώρα. Το ίδιο ισχύει και για τα τύρανα. Ε, Τώρα η διαδικασία γίνεται πιο σύνθετη. Στο βαθμό που οι, μετα... οι μεταρρυθμίσεις και ενταξιακή διαδικασία γίνονται εκ παραλίλου, δεν χρειάζεται να υπάρχει μια συνένεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη προοπτική η οποία να μετατρέπεται σε πράξη πριν είναι υπερβολικά αργά γιατί υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι έχουν βλέψει στην περιοχή παρόλο που δεν είναι συμβατές με τις ευρωπαϊκές αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει την αξιοπιστία της παγκοσμίω, δίνοντας ένα θετικό παράδειγμα στην άμεση γειτονία της και στη συνέχεια και αλλού. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο, κύριο Σεζουνέ. Είμαι υπέρ τη διεύρυνση. Είμαι υπέρ του αυτέ οι δύο χώρε να μπορέσουν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, πώς μπορούμε να προσθέσουμε άλλες δύο έδρε στο Συμβούλιο σήμερα, παρόλο που τα θεσμικά μας, ε, το θεσμικό σύστημα ε, είναι σε αδιάξοδο. Εγώ πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα δεν είναι αιώνια, θα πρέπει να τα προστατεύσουμε και θα πρέπει σε κάποια συγκυρία να ε, θέσουμε το ερώτημα της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο πριν θέσουμε την, το ζήτημα της διεύρυνσης. Εγώ είμαι ευρωπαϊστής και πραγματικά αναλαμβάνω την ευθύνη αυτής της ε, θέσης. Ε, θα πρέπει να θέσουμε το ζήτημα της αναθεώρησης του Συμβουλίου πριν θέσουμε το ζήτημα της προσθήκης δύο ευρών εδρών στο Συμβούλιο. Νομίζω θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να σκεφτούμε την Ευρώπη σε 10-20 χρόνια. Εγώ είμαι ευρωπαϊστής και δεν θα, δεν θα ήθελα να ισχύσουμε τον αντιευρωπαϊσμό ε, ε, δημιουργώντας νέα προβλήματα λοιπούς ε, αποτελεσματικότητας. υπόσχεση προς Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία και να ενισχύσει την σταθερότητα και την ειρήνη στα Βαλκάνια. Αντίθετα, κατάφερε ισχυρό πλήγμα στους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων. Η απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και είναι σαφέ ότι οι χώρε θα πληρούν. Η Γαλλία και η Ολλανδία όμω ε, ε, φέρθηκαν ανεύθυνα, αλλάζοντα στη μέση του παιχνιδιού του κανόνε. Έτσι, οι πολιτικές, ε, πολιτικές σκέψεις αυθαίρετες τώρα επηρεάζουν τους λαούς και τις κυβερνήσεις των δύο χωρών που έκαναν τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις. Η απόφαση είναι μειοντική. Ε, δημιουργεί κινδύνους μακροπρόθεσμα για όλη την περιοχή. Το μήνυμα του Συμβουλίου και του Μακρόν είναι ότι δεν θέλουν να πληρούν τα κριτήρια ανεξάρτητα από τις προσπάθειες. Εμείς θα συνεχίσουμε να τους ε, ενθαρρύνουμε και να τους θυμίζουμε ότι τα θεσμικά όργανα και τα περισσότερα κράτη-μέλη θέλουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις και το Συμβούλιο πρέπει να το δείξει αυτό ε, ανατρέποντας την ε, αρνητική απόφαση το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και τι δεν θα κάναμε για χώρες τις οποίες η μερίσια ή ε, όχι, η μηνιαία αμοιβή δεν ξεπερνάει τα 400 ευρώ ο μηνιαίος μισθός. Βλέπουμε λοιπόν ότι το οικονομικό κριτήριο ε, ακυρώνει μερικές φορές τις ατέλειες μιας χώρας όπως η Αλβανία με παρουσία του ριζοσπαστικού Ισλάμ και με ε, πολλούς τζιχαντιστές ε, με το τέμενος του Ναμαζγκά που χρηματοδοτείται από την Τουρκία και δείχνει την κυριαρχία του Ερντογάν, μια χώρα με λαθρεμπόριο από παντού, ε, με υψηλότατο δίκτυ στην κατάταξη της διαφθοράς στην Ευρώπη και στην Βόρεια Μακεδονία η ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή για τη Συμφωνία των Πρεσπών και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει την αλήθεια. Ας κλείσουμε λοιπόν το κεφάλαιο της διεύρυνσης και των εκατομμυρίων ευρώ που σκανδαλωδώς σπαταλάμε ε, στα πλαίσια της προένταξης. Κοιτάξτε, πριν περάσουμε στον επόμενο μιλητή, θα ήθελα να καλωσορίσω στους επισκέπτες της Ολομέλειας. Έχουμε τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βόρειας Μακεδονίας, τον αξιότιμο κύριο Ταλάτ Τσαφέρη και τον καλωσορίζουμε. Ε, σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην συζήτηση αυτή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Εύχομαι οι συναντήσεις σας να είχαν ενδιαφέρον. Περνάμε λοιπόν συναδελφοί τώρα στον επόμενο ομιλητή, ο κύριος Τομασεύσκη για ένα λεπτό. Okay, I don't think the... δεν νομίζω ότι είναι στην αίθουσα ο ομιλητής. Προχωρούμε. 1,5 λεπτό. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Υπάρχει μια αλλαγή στον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Η έλλειψη απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ε, για αναβολή για μια ακόμη φορά της έναρξης των διαπραγματεύσεων είναι ιστορική εμβέλειας λάθος. Ε, είναι κάτι που αγνοεί τις θέσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αγνοεί τις δικές μας θέσεις, αγνοεί τις επιθυμίες των εταίρων μας, που όλοι διαιρωτώνται ε, για τις πραγματικές μας επιθυμίες. Η Αλβανία και ιδιαίτερα η Βόρεια Μακεδονία έκαναν πολλές προσπάθειες. Άλλαξε και το όνομά της η χώρα αυτή για να υπογράψει μια ιστορική συμφωνία με την Ελλάδα. Δυστυχώς η αξιοπιστία μας κλονίστηκε. Είχαμε πει ότι θα αξιολογήσουμε τις επιδόσεις τους με αντικειμενικό τρόπο. Αυτό δημιουργεί ένα ανησυχητικό προηγούμενο και ανοίγει τις πόρτες των Βαλκανίων στους ανταγωνιστές μας. Ο Ερντογάν επισκέπτεται τη Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία πέφτει σε μια σοβαρή πολιτική κρίση. Λέω στους φίλους από τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία καλό κουράγιο, θάρρος και δεν θα σταματήσουμε ε, μέχρι ότου ανατρέψουμε την απόφαση του Συμβουλίου. Ο κύριος Μπίλτσικ, ένα μισή λεπτό. Η απόφαση της περασμένης εβδομάδας του Συμβουλίου κλώνησε τα θεμέλια μιας πιο πολύ επιτυχούς πολιτικής. Τώρα ε, έχουμε ένα ανοιχτό γεωπολιτικό πρόβλημα χάρη της ομοφωνίας. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις δύο χώρες ε, ε, θα έπρεπε να αρχίσει. Η αποτυχία αυτή είναι από τα μεγαλύτερα σφάλματα. Είναι προς το αμοιβαίο και κοινό συμφέρον να προχωρήσουμε προς την ένταξη. Υπάρχουν χώρες ε, που απορρίπτουν την διεύρυνση. Αν θέλουμε όμως ισχυρή ένωση, διεθνώς σεβαστή, θα πρέπει να έχουμε αποφασιστική φωνή και να σκούμε επιρροή στην άμεση γειτονία μας. Η απογοήτευση σήμερα στα Δυτικά Βαλκάνια είναι τεράστια. Η Βόρεια Μακεδονία άλλαξε το όνομα της χώρας για να πάρει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση οδήγησε σε ενοποίηση και αίσθηση ασφάλειας στην, ε, στα Βαλκάνια. Αυτό όμως δεν είναι δεδομένο ε, πάντοτε, ιδιαίτερα βλέποντας τη δράση της Τουρκίας στη γειτονιά μας. Χρειαζόμαστε ε, ανθεκτική, δημοκρατική, ανθεκτικά, δημοκρατικά, ειρηνικά Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό θα είναι και δική μας επιτυχία. Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σάντος, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη και γνωρίζω ότι την απογοήτευσή μου τη σημερίζω δηλαδή της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας γιατί βλέπουν ότι το όραμά τους να ε, προσχωρήσουν στην Ένωση ε, αποκλείστηκε μετά τις ε, μετά το βέτο ε, της ε, Γαλλίας και οι δύο χώρες παρά τις προτάσεις ε, της Κομισιόν και οι δύο χώρες πληρούσαν τα κριτήρια και προχώρησαν στις μεταρρυθμίσεις που τους ζητήσαμε. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να σταματήσει. Κι όμως το Συμβούλιο ε, ε, έπεσε όμοιρο στα χέρια του κυρίου Μακρόν και άνοιξε και το ενδεχόμενο και άλλοι παίκτες να ασκήσουν επιρροή σε αυτήν την σημαντική για την Ευρώπη περιοχή. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση φανεί ανίκανη να έχει ένα στρατηγικό όραμα και να αναλάβει ηγετικό ρόλο, δεν θα θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Και προχωρούμε προς ε, πλήρη απαξίωση. Το Συμβούλιο απέτυχε, αλλά εδώ εμείς στο Κοινοβούλιο συνεχίζουμε τη μάχη για να τηρηθούν οι υποσχέσεις μας. Ένα λεπτό ο κύριος Γκροσέλτσε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λυπούμε για την απόφαση του Συμβουλίου να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες και απογοητεύομαι διότι δεν αναγνώρισε τις, ε, τους συμβιβασμούς που έπρεπε να κάνουν οι δύο χώρες καθοδόν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η... Ακούω για μεταρρύθμιση της διαδικασίας ε, ε, ένταξης πριν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Όμως αυτό δεν είναι εμπόδιο αν υπάρχει αρκετή πολιτική βούληση. Εμείς θέλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή θεσμικά δεν μπορεί να στηρίξει χώρες που δεσμεύονται υπέρ των δημοκρατικών αξιών. Είναι τελείως λάθος μήνυμα να αποστέλουμε, αυτό το μήνυμα που αποστέλουμε στι, στις γειτονικέ χώρες. Αυτό ισχύει κυρίως για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου η, δυτική, ε, όπου η Βόρεια ε, ε, Μακεδονία είναι μια χώρα όπου υπάρχει αύξηση του λαϊκισμού. Ε, θα υπήρχε ε, η δυνατότητα να στείλουμε μήνυμα ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Οι χώρες που απορρίπτουν τον λαϊκισμό, τη διαφθορά έχουν ε, ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Αν δεν μπορούμε να το στείλουμε, να το πούμε σαφώς. Μην ξεπερνάτε το χρόνο γιατί ήδη είμαστε σε καθυστέρηση και θα σας διακόψω κλείνοντας το μικρόφωνο αν δεν τηρήσετε το χρόνο σας. Κύριε Πρόεδρε, αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις. Την αβεβαιότητα του Brexit. Γιατί λοιπόν πρέπει σε αυτή τη συγκυρία να σκεφτούμε σοβαρά να προσχωρήσουν η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία στην Ευρώπη και στις δύο χώρες η ανεργία είναι υψηλή, η μισθή είναι χαμηλή ε, δεν και υπάρχουν τεράστια ελλείμματα. 60% ε, των ενήλικων στην Αλβανία επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Άρα λοιπόν υπάρχουν εύλογες ε, Ανησυχίε ε, και σε μια, πόσο μάλλον σε μια συγκυρία που ήδη οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν ε, μεγάλα προβλήματα. Οι συνεχείς προσπάθειες για διεύρυνση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πάντοτε θετικές. Ας διακόψουμε τις, ε, τη διαδικασία ένταξης και ας σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνδράμουμε τις χώρες μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και να επιστρέφοντας σε μια ισορροπημένη πολιτική προκειμένου να ενισχύσουμε χώρες αυτές και να διακόψουμε την επιρροή τρίτων χωρών. Ο κύριος Ρτζόγκα, ε, κυρία, κυρίες και κύριοι, κύριε Πέτροπε, η, το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέστη ένα σοβαρό πλήγμα. Ε, ήταν μια απόδειξη ότι τα συμφέροντα της Γαλλίας έχουν ε, προτεραιότητα εναντί των ε, συμφερόντων του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Βόρεια Μακεδονία εκπλήρωσε όλα τα κριτήρια και αυτό το γνώριζαν όλοι οι πολίτες της χώρας. Γι' αυτό θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο αυτό εξετέθη ε, ε, σοβαρά. Ε, δεν είναι καλό αυτό για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε για την ευρύτερη περιοχή. Η Βόρεια Μακεδονία ε, στη χώρα αυτή μάλλον της άνοιξε ο δρόμος για το ΝΑΤΟ. Η Βόρεια Μακεδονία έκανε πολλές προσπάθειες για να πετύχει αυτό το στόχο. Ίσως πρόκειται για την επιβολή αντιπίνων. Η κυρία Φοντερ Λάιν ήταν υπέρ της διεύρυνσης, αλλά ο υποψήφιος του Μακρόν δεν πέρασε την ακρόαση στο Κοινοβούλιο και ίσως αυτά ήταν τα αντίπινα. Ο κύριος Σανλαβάνος για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Τα βάσανα από τα οποία έχουν υποφέρει οι λαοί των βαλκανίων έχουν συγκεκριμένε αιτίε. Αυτέ είναι οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οι νατοικές επεμβάσει οι αλλαγέ των συνόρων οι ξένες στρατιωτικές βάσεις η υποκίνηση των εθνικισμών η διασύνδεσή του με την ευρωπαϊκή ένωση οι καπιταλιστικέ αναδιαρθρώσεις. η εμπειρία αποδεικνύει ότι καμία ένταξη χωρών στην ευρωπαϊκή ένωση και το νάτο δεν μπορεί να γίνει προ όφελο του λαού. αντίθετα αυτή υπαγορεύεται από τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. εκεί ακριβώς οφείλεται και η αντιπαράθεση που γίνεται εντός της ευρωπαϊκής ένωσης για την ένταξη της βόρειας μακεδονίας δηλαδή στους οξύς ανταγωνισμούς της γαλλίας της γερμανίας άλλων χωρών για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στα δυτικά βαλκάνια στο φόντο της σκληρής πολιτικής οικονομικής σύγκρουσης της ευρωπαϊκής ένωσης των ηνωμένων πολιτειών του νάτο με τη ρωσία και την κίνα στην περιοχή. οι αντιπαραθέσει μεταξύ των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης δεν αμφισβητούν την επιζήμια για τους λαούς συμφωνία των πρεσπών ευρωνατοικής σκοπής που υπογράφηκε με στόχο την ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή ένωση και στο νάτο. οι λαοί των δυτικών βαλκανίων αλλά και ολόκληρης της ευρώπης μπορούν να ζήσουν ειρηνικά έξω όμως από τον κορσέ της ευρωπαϊκής ένωσης έξω από το νάτο από τον κορσέ των υπεριαλιστικών σχεδιασμών απορρίπτοντας τον εθνικισμό τον αλυτρωτισμό με την εξουσία και την οικονομία στα δικά τους χέρια. Κύριε δεν είναι ανάγκη, δεν να αναφέρομαι και πάλι ότι ήταν λάθος και πολύ κακή απόφαση. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο σημαντικό ήταν για, όλο, για όλη την Ήπειρο και είναι και θα είναι και στο μέλλον η πολιτική διεύρυνση της Ένωσης. Ούτε χρειάζεται να επαναλάβουμε πόσα πολλά πράγματα έγιναν, πόσες επώδυνες ε, μεταρρυθμίσεις έγιναν, ε, κυρίως από τη Βόρεια Μακεδονία αλλά και την Αλβανία και πόσο νιώθουν σήμερα ε, ότι έχουν εξαπατηθεί από εμάς. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα είναι πολύ απλό. Τι πρέπει να αλλάξουμε από τη δική μας την πλευρά, από την πλευρά της Ένωσης, ούτως ώστε η διαδικασία διεύρυνση να μην μπλοκαριστεί από ένα κράτος μέλος. Τι μπορεί να αλλάξει. Πριν προχωρήσουμε στις ε, μεταρρυθμίσεις για την ένταξη, θα πρέπει να ε, έχουμε έναν απλό κανόνα. Να ζητήσουμε από τις χώρες που μπλοκάρουν τις αποφάσεις του Συμβούλιο να έρχονται εδώ και να μας εξηγούν τα επιχειρήματά τους. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα επιχειρήματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορεί έτσι να βρούμε έναν τρόπο για να πείσουμε τα κράτη-μέλη να ξεπεράσουν την άρνησή τους. Πρέπει λοιπόν να μας απασχολεί όχι μόνο η υποστήριξη στις δύο χώρες που την αξίζουν, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε και τη Γαλλία να ξεπεράσει το λάθος της. Γιατί αυτό δεν είναι λάθος μόνο της Γαλλίας, αλλά ουσιαστικά είναι λάθος όλων μας. Ευχαριστώ κύριο Σίντερ ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε πολύ σωστά ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση κύριος Χάν, η απόφαση είναι βαρύ λάθος και την ευθύνη την φέρει στο Συμβούλιο ο, Γαλλικό, ο Γάλλος Πρόεδρος. Όμως οι επιπτώσεις αυτού του σφάλματος θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από όλους εμάς στην Ευρώπη, ε, από όλους μαζί. Ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρεί τις υποσχέσεις που έκανε προς την ε, Βόρεια ε, Μακεδονία και την Αλβανία που έκαναν τόσο σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα η Βόρεια Μακεδονία έλυσε το θέμα του ονόματος και τα προβλήματα με τη γείτονα χώρα. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ε, διορθώσει το λάθος το ταχύτερο δυνατόν. Αλλά και εμεί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία μέσω διμερών διαπραγματεύσεων, μέσω της ε, ε, διαδικασίας αμονή να Έχουμε πιο στενές επαφές με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και να τους δείξουμε ότι την απόφαση θεωρούμε λάθος και ότι ελπίζουμε να διορθωθεί σύντομα. Ο κύριος Πάετ, ένα λεπτό. Ευχαριστούμε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει μια νέα και στρατηγική απόφαση, γιατί ήταν σφάλμα να μην, αρχίσει, να μην υπάρξει έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Η προοπτική προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κινητήρια δύναμη για τι αλλαγέ που έγιναν στι δύο αυτέ χώρε. Η Βόρεια Μακεδονία οδηγήθηκε να πιστέψει ότι αλλάζοντα το όνομα θα μπορέσει να προχωρήσει προσεγγίζοντα περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, Βεβαίω, οι μεταρρυθμίσει στην πραγματικότητα θα πρέπει να γίνονται για, την, για εσωτερικούς λόγους. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ξεκινήσει τις ενταξιακές δραπαγματεύσεις και με τις δύο χώρες προκειμένου να τις ενθαρρύνει για να συνεχίσουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες και, να έχουν, και προκειμένου και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αξιόπιστους εταίρους. Ωστόσο, Επίσης ε, υπάρχει και η δυνατότητα άσκησης επιρροή στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών ε, Βαλκανίων. Είναι δύσκολο να φανταστούμε να επιτυχαίνει στο ρόλο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν ε, αστόχησε στην προσπάθεια ένταξη των χωρών αυτών. Ο κύριος, η κυρία Χουτασάρη, το καθεστώ της υποψηφία προ ένταξη χώρας έπρεπε να δίνεται μόνο σε χώρε που έχουν πραγματικές πιθανότητες να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο αυτές χώρες πλήττονται από το έγκλημα και έχουν υψηλά ποσοστά διαφθοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη σοβαρά προβλήματα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 ενώ δεν ήταν ακόμη έτοιμες. Δεν θα πρέπει να δίνουμε ψεύτικες ελπίδες σε χώρες που στην πραγματικότητα δεν εκπληρούν τα κριτήρια να γίνουν υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάψει να διευρύνει τα σύνορά της όταν δεν μπορεί να διευθετήσει τα του οίκου της. Mr. Lagos. Ο κύριος Λαγός για 1,5 λεπτό. Πριν από λίγο από κάποιους ομιλητές ότι υπήρξε μεγάλο πολιτικό θάρρος για να φτάσουμε στη συμφωνία των σκοπίων ε, με την πατρίδα μου την ελλάδα. θα ήθελα να πω μέσα σε αυτή την αίθουσα για να ακουστεί ότι δεν υπήρξε κάποιο πολιτικό θάρρο, ξέρετε αλλά υπήρξε η επιβολή πραγματικά μια μικρή μειοψηφία, ει βάρο της θέλησης του ελληνικού λαού. πάνω από 75% των ελλήνων έω 80% δεν ήθελαν με τίποτα τη συμφωνία αυτή. Στι απαιτήσει των ελλήνων για να γίνει δημοψήφισμα η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε κατηγορηματικά. έτσι φτάσαμε λοιπόν η κυβέρνηση τότε και η σημερινή κυβέρνηση να είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτέ αυτή τη προδοτική συμφωνία που έχει γίνει ει βάρο τη πατρίδα μα. και όσο αφορά όλου του ευρωβουλευτέ εδώ αλλά και του κατοίκου όλων των ευρωπαϊκών χωρών πρέπει να βγουν από την πλάνη αυτή. δεν υπάρχει βόρεια μακεδονία υπάρχει το κράτο των σκοπίων για να το ξεκαθαρίσουμε. το ξέρουν όλοι οι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν είναι λόγια που λέω εγώ ή κάποιοι έλληνε εθνικιστέ. και όσο αφορά για να το κλείσουμε και για να γίνει σαφέστατο όλο αυτό εδώ υπάρχει αναγραφόμενη σε μια μαρμάρινη πλάκα που είχε βρεθεί πριν από λίγο καιρό στην πατρίδα μου μια επιγραφή. Η επιγραφή αυτή λέει Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν. Η επιγραφή αυτή, εγώ που είμαι Έλληνα, ξέρω και τη διαβάζω μετά από δύο, χιλιάδε χιλιάδες χρόνια. Οποιοδήποτε κάτοικο των Σκοπίων δεν μπορεί να διαβάσει αυτή την επιγραφή. Άρα μη σου πράγματα που δεν του ανήκουν. Η Μακεδονία είναι μόνο μία και είναι μόνο ελληνική. σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε επίτροπε χαν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών βαλκανίων οφείλει να παραμείνει ανοιχτή και διότι λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή και γιατί αποτελεί δημοκρατικό μοχλό πίεσης για τον απαραίτητο εξυγχρονισμό των χωρών αυτών είναι επίσης απαραίτητο οι κυβερνήσεις στα τύρανα και τα σκόπια να γνωρίζουν ότι δεν αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων σε σχέση με τις χώρες που προηγήθηκαν. ειδικά η αλβανία οφείλει να σέβεται την ελληνική μειονότητα και τα δικαιώματά της. αντίθετα έχουμε επανειλημμένες παραβιάσεις τα τελευταία χρόνια. σε ό,τι αφορά τη βόρεια μακεδονία στηρίζουμε την ευρωπαϊκή της προοπτική. η προηγούμενη κυβέρνηση μέσω της συμφωνίας των πρεσπών αποδέχθηκε τη σύνδεση της εφαρμογής της σύνθετης ονομασίας έναντι όλων έργα omnes με το άνοιγμα των κεφαλαίων κατά την ενταξιακή πορεία. η ενταξιακή πορεία είναι εκ των πραγμάτων απαραίτητη για την ύπαρξη της σύνθετης ονομασίας έναντι όλων που αποτέλεσε και το διαβατήριο της χώρας αυτής για τον νατο. σας ευχαριστώ. κύριε Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η αναποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας στέλνει τελείως λάθος μήνυμα στους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων και όχι μόνο τους ε, κατοίκους της Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας. Και το πιο λάθος μήνυμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τύχει εμπιστοσύνη. Όσες προσπάθειες και θυσίες κάνεις μπορεί να σε εξαπατήσουν. Και μάλιστα, όχι για σοβαρό λόγο, αλλά για τις δημοσκοπήσεις, χάρη των δημοσκοπήσεων σε μια χώρα. Η επιρροή της Ένωσης ως περιφερειακός παίκτη ε, θα αρχίσει να δει, παρόλο που τα πράγματα συνεχίσουν, ο ήλιος θα συνεχίσει να ανατέλει στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Εμεί περιμένουμε τι μεγαλειώδει ευρωπαϊκέ μεταρρυθμίσει που θέλει ο κύριο Μακρόν. Άλλοι όμω ε, θα είναι ευτυχεί να καλύψουν το κενό που αφήνουμε εμεί. Ε, δεν θα ανανεώσουμε την Ευρώπη αθετώντας τις υποχρεώσεις μας και τις υποσχέσεις μας και κάνοντας βασικές ενωσιακές πολιτικές όμοιρο σε, εγωιστικές, σε εγωιστικά συμφέροντα. Αυτό ενισχύει τον λαϊκισμό και τον εθνικισμό. Ο κύριος ε, Σίμετσκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους ε, που είπαν ότι η αναποφασιστικότητα του Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα ήταν μεγάλο στρατηγικό σφάλμα. Και το πρόβλημα τώρα είναι ότι η αξιοπιστία της ε, Ευρώπης διεθνώς έχει ζημιωθεί. Εμείς ε, ισχυριζόμεθα ότι είμαστε οι ε, ε, αμύντορες των αξιών μας, αλλά δεν ανταποκριθήκαμε στους κανόνες που θέσαμε για τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε μερεσιμότητα βάσει σαφών αντικειμενικών κριτηρίων και οι συζή... μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα τα βελτιώσουμε αυτά, αλλά δεν μπορούμε ε, να ε, αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Και αυτό ε, βλέπουμε πόσο ζημιογόνο ήταν και βλέποντας την πολιτική κρίση στη Βόρεια Μακεδονία και τα προβλήματα στην Αλβανία. Δεν πρέπει να σταματήσουμε την ε, διεύρυνση, επειδή μπορεί να υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με το κράτος δικαίου σε κάποιες χώρες. Θα πρέπει αντίθετα να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Ο κύριος Μπαρντέλα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συζητάμε την πιθανότητα η Αλβανία να γίνει μέλος της Ένωσης. Μια χώρα η οποία de facto είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Αλβανοί υπάρχουν στην Γαλλία μου ας πούμε και α, μέσω μαφιόζικων οργανώσεων κυκλοφορούν ελεύθερα με παράνομες δραστηριότητες. Το να ανοίξουμε τις πόρτες στην Αλβανία θα επιτείνει μια κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη το σύνολο των ε, λαών της Ευρώπης θέλουν να προστατεύσουν την ταυτότητά τους και τον τρόπο ζωής τους και τους προτείνουμε μια χώρα η οποία έχει απόμακρες αξίες και επηρεάζεται άμεσα από την Τουρκία του Εντοάν. Με τις τελευταίες ευρωεκλογές έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα οι λαοί της Ευρώπης. Ε, όρια στις τράπεζες, όρια ε, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ε, βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει παραλύσει ενώ όλες οι άλλες περιοχές του κόσμου ευημερούν. Μπλε κάρτα, δέχεστε την ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διερωτώ με πότε επισκέφτηκε τα Τύρανα, το μοναστήρι, τα Σκόπια. Ε, είναι μια παράλογη συζήτηση. Κάποιες χώρες θέλουν να μπουν στην Ένωση θέλουν να μπουν και κάποιες που είναι στην Ένωση θέλουν να βγουν. Κοιτάξτε, πρέπει να τελειώνει αυτή η συζήτηση. Όταν έχεις υποσχεθεί κάτι σε κάποιον πρέπει να τηρήσεις την υπόσχεσή σου γιατί την επόμενη φορά δεν πρόκειται να σου δείξει εμπιστοσύνη. Είναι ιστορικό το λάθος, στην ουσία εδώ παίζουμε με την ειρήνη και η ερώτησή μου ε, πώς μπορούν να ζήσουν με διαφορετικό τρόπο οι άνθρωποι αυτοί αν δεν γίνουν μέλη της Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ εκλέγομαι στη Γαλλία και προασπίζομαι τα συμφέροντα του γαλλικού λαού. με απασχολεί η ευημερία του λαού μου. Εσείς προτιμάτε να προστατεύσετε την ευημερία των άλλων και όχι των δικών σας. Αλλά οι λαοί της Ευρώπης εξεφράστησαν μαζικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκλογών. Οι λαοί της Ευρώπης θέλουν την προστασία της ταυτότητάς τους, θέλουν την προστασία της ε, κυριαρχίας τους, της δημοκρατίας τους. Και δυστυχώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστεί ακριβώς τα αντίθετα. Ο κύριος Ραντατσόφσκι 1,5 λεπτό. οι χώρες αυτές έλαβαν ένα ράπισμα, ισχυρό ράπισμα στο πρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν θα, δεν θα ανοίξουν οι ενταξιακές πραγματεύσεις. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πάντα. Ε, θέλουν η, Μακεδονία να μπει, ε, είπαμε στη Μακεδονία να μπει στο ΝΑΤΟ για να παίξει το παιχνίδι των Αμερικάνων. Δώσαμε υποσχέσει ε, στην Αλβανία και δεν τις εκπληρώσαμε. Τα αμερικανικά ελικόπτερα μπορούν τώρα να προσγειωθούν στην Μακεδονία, στη Βόρεια Μακεδονία γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα να δεχτείτε στην Ευρώπη ε, μικρές ε, χριστιανικές ε, χώρες τις οποίες αντιμετωπίζετε σαν να είναι ε, κατηγορίες σαν να είναι δευτέρας κατηγορίας χώρες. Mr. Ο κύριος Μπρέσλερ, ένα λεπτό. Η πολιτική της διεύρυνσης είναι από τις πιο πετυχημένες ενωσιακές πολιτικές. Ένωσε την Ευρώπη, έφερε σταθερότητα, ασφάλεια. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο να μπλοκάρουμε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ε, ε, πόσο μάλλον που υπήρχε θετική σύσταση από την Κομισιόν με βάση τα επιτεύγματα. Θα πρέπει οι υποψήφιες χώρες να αξιολογούνται αποκλειστικά με βάση τα αποτελέσματα και όχι να επηρεάζονται από καταστάσεις ε, σε άλλα κράτη-μέλη. Ας είναι και μεγάλα κράτη-μέλη. Αυτό το τεράστιο ιστορικό σφάλμα θα ενισχύσει τους άλλους παγκόσμιους παίκτες στην περιοχή. Και αυτή η ανευθυνότητα θα αμφισβητήσει επίσης την αξιοπιστία της Ένωσης. Γι' αυτό η σύνοδος στο Ζάγκρεπ το Μάιο του χρόνου θα είναι μια ευκαιρία να εστιάσουμε σε αυτή την περιοχή και να θέσουμε σαφείς ε, καταληκτικές ημερομηνίες. Ε, ευχαριστώ ε, κύριε ε, Πρόεδρε. Οι νέοι χάνουν την ελπίδα τους στην, ε, στα Βαλκάνια. Δεν μας εμπιστεύονται, δεν μας πιστεύουν και δικαίως. Να θυμίσω τα λόγια του Γάλλου Προέδρου το περασμένο φθινόπωρο που είπε πριν από το ε, δημοψήφισμα για τις πρέσβες υπολογίζουμε σε εσά και είναι ο ίδιος πρόεδρος ο κύριος Μακρόν τον οποίο ρωτώ θα αναλάβει ευθύνη για τη σταθερότητα στην περιοχή, θα αναλάβει ευθύνη για τις πρόορες εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία. Οι κενές υποσχέσεις ε, είναι το μόνο που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλάμε για τη διεύρυνση, που είναι πισόπλατη μαχαιριά στους λαούς ε, της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας και των Βαλκανίων. Εδώ και δέκα χρόνια ε, ε, έπαιρνε υποσχέσεις ε, η Βόρεια Μακεδονία ότι αν έκανε κάποια βήματα θα άρχιζε διαπραγματεύσεις. Είναι κρίμα. Πρέπει να δείξουμε πνεύμα υπευθυνότητας και να συζητήσουμε τι απόφαση θα πάρουμε για τη διεύρυνση στο μέλλον. Να διορθώσουμε επίσης τα σφάλμα μας από αύριο. Ευχαριστώ. Ήθελα να αντιδράσω σε είπε η κυρία Φαγιόν, διότι θα πρέπει να δείξουμε την ίδια αξιοπιστία και να επιτρέψουμε την προσχώρηση στο χώρο του Σέγγεν, αφού δώσει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,